τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα ώστε να υπάρχει ισοτιμία ε, στις εμπορικές συνδιαλλαγές και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των μισθωτών. Σας ευχαριστούμε κύριε Νά. Ε, η κυρία